Οι αρμόδιες αρχές ε, της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας μου γνωστοποίησαν την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των ε, Γύρι Πάινε, Ρατσβαν Πόπα, Ασίμα Μαχμέντοφ Αντέμοφ και Λίβια Γιαρόκα από τις 5, 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2017 αντιστοίχως και αντικαθιστούν αντιστοίχω τους Μάκα, Νεγκρέσκου, Γκάμπριελ, Γκαλπέλτσε. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση τη εντολής του. καλωσορίζω τους νέους συναδέλφους και υπενθυμίζω ότι συμμετέχουν με πλήρη δικαιώματα στο Κοινοβούλιο και στα οργανά του υπό τι προποθέσει προβλέπονται στον κανονισμό.